Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε στην κοινή αυτή συνεδρίαση των Επιτροπών Εξωτερικών και Ανάπτυξης για μια ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο Τάμπου Μπέκη, που είναι πρόεδρος της Υψηλής Επιτροπής του Ψηλού Πάνελ για τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Χαίρομαι πολύ. Σας γνώρισα και ως αντιπρόεδρο και ως πρόεδρο. Σήμερα έχετε να ε, μας ενημερώσετε, όχι να επιλύσετε, ελπίζουμε βέβαια να γίνει και αυτό, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι και ο Δ. Αμπτουλάη και ο Δόκτωρ Χάντοκ και άλλα μέλη του πάνελ. Πριν από δύο χρόνια, κύριε Πρόεδρε, είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Είστε εδώ σήμερα για να μα παρουσιάσετε τα απορίσματα της τελικής έκθεσης του πάνελ που εκρήθηκε ε, την προηγούμενη χρονιά. Δίνει πραγματικά μας ε, κάποια ανησυχητικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως είναι για πόλεις ε, για την ε, Αφρικανική Ήπειρο. Και όλα αυτά βέβαια καταδεικνύουν πόσο αναγκαίο είναι να ληφθεί δράση και σε διεθνές παγκόσμια αλλά και σε τοπικό επίπεδο. παράνομες χρηματοοικονομικές ροέ απειλούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια των αφρικανικών χωρών υπονομεύουν τους θεσμούς, στη δημοκρατία, θέτουν σε κίνδυνο την βιώσιμη ανάπτυξη και το κράτος δικαίου. Επίσης, είναι ζητήματα που ανησυχούν σοβαρά και έναν από τους σημαντικούς παρόχους της χρηματοοικονομικής βοήθειας και ενίσχυσης προς την Αφρική της ΕΠΑ. Μιλάμε τώρα βέβαια και για τη μετανάστευση και πολλά μας ανησυχούν. Έχουμε τη Λιβύη, τόσους πολλούς ανθρώπους που ναυαγούν και χάνουν τη ζωή τους και σίγουρα θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει ζωές ε, αν τα χρήματα εκεί ε, χρησιμοποιούνταν για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου στην Αφρική. Οπότε θα ήταν λιγότεροι μετανάστες και λιγότεροι και οι νεκροί στη Μεσόγειο. Να δούμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Στην έκθεση διατυπώνονται ορισμένες σημαντικές στάσεις ε, και περιμένουμε ανυπομονησία. Να ακούσω από εσάς πώς θα μπορούσε να ε, υλοποιηθούν, πώς θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και πώς θα μπορούσε να βοηθήσει και το Κοινοβούλιο. Να σας υπενθυμίσω τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να ενισχύσει τις διατάξεις για τη δέωση επιμέλεια σε ό,τι αφορά παραδείγματο χάρη ε, τα μεταλλεύματα από εμπόλεμες περιοχές, για τη βελτίωση της ε, διαφάνειας και τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε ό,τι αφορά αυτές τις βασικές πρώτες ύλες. Ε, πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ επίκαιρο και έγκαιρο. Έχουμε την αποκάλυψη των γράφων του Παναμά. Βλέπουμε να υπάρχουν σχετικά ε, διασυνδέσεις. Θα δώσω τώρα το λόγο στην συνάδελφο Μακάβα. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Μπέκη, καλώς ορίσατε ε, στην ε, κοινή αυτή συνεδρίαση των Επιτροπών Άφρικ και Ντέβη για τη δική μου Επιτροπή, την Επιτροπή Ανάπτυξης, η οποία είναι αρμόδια με επιβλέπει τις πολιτικές για την ανθρωπιστική βοήθεια, την αναπτυξιακή πολιτική, σίγουρα η αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών αποτελεί προτεραιότητα. Όπως είπε και ο Έλμαρ Μπρόκαν, τα χρήματα αυτά δίνονταν, ήταν διαθέσιμε σε ανεπτυσσόμενε χώρε, θα έκαναν τεράστια διαφορά στι ζωέ αυτών των ανθρώπων. Μιλούμε για του βιώσιμου ε, αναπτυξιακού στόχου. Ε, πέρυσι στη Νέα Υόρκη, όπου συγκεντρώθηκαν ηγέτε, ε, είπαν πολλά και καλά λόγια. Είπαν για την παγκόσμια περίθαλψη και υγεία, για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, τη τα κτλ. Ωραία λόγια που όμω δεν σημαίνουν τίποτε εάν δεν αντιμετωπίσουμε στην πράξη αυτά τα προβλήματα. Είπε και ο ε, ότι είχαμε τις αποκαλύψεις ε, των εγγράφων του Παναμά που έριξαν φως στην κατάσταση αυτή. Είναι κάτι που δεν μπορούν να το δεχτούν οι πολίτες πια ούτε στην Αφρική ούτε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας νόμος για τους πλουσίους και άλλος νόμος να ισχύει για τους υπολείπους. Ε, μόνο αν πληρώνουν όλοι τους φόρους τους μπορεί να υπάρχει μια αξιοπρεπής κοινωνία, μπορούν να, τα κράτη να λειτουργούν και να μην χάνονται τα κρατικά έσοδα. Πολλές εταιρείε μπορούσαν καν ε, να έχουν κέρδος αν δεν είχαν επενδύσει στην εκπαίδευση, στις υποδομές, στο δικό δίκτυο κτλ. οι κυβερνήσεις. Ε, πέρυσι η Επιτροπή μας, η γνώμη, με την συνάδελφο Έντι Λάιν συγκεκριμένα ε, συνέταξε μια έκθεση για το θέμα αυτό και στην που το συζητήσαμε στη σχετική διάσκεψη και θα θέλαμε να συνεργαστούμε και μαζί σας για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που απαιτούν μια ευρωπαϊκή αλλά και μια παγκόσμια προσέγγιση. Σας καλωσορίζω θερμά σήμερα εδώ και είναι καλό που συναντούμε και την ομάδα σας να δούμε πώς μπορούμε στο μέλλον να, να ε, συνεργαστούμε ακόμη πιο αποτελεσματικά. Κύριε Μπέκη, έχετε το λόγο. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπρόεδροι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να συζητήσουμε μαζί σας το ζήτημα αυτό των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών από την Αφρική. Όπως άλλο τυπώθηκε, ήμασταν ε, εδώ και πριν από ορισμένα χρόνια προκειμένου να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό και προκειμένου να καταλήξουμε σε μια κοινή κατανόηση για το τι θα μπορούσε να γίνει για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Προετοιμάσαμε μάλιστα και μία έκθεση, στα πλαίσια της οποίας προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με πάρα πολλές κυβερνήσεις από την Αφρική, με διάφορους διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και προσπαθήσαμε ουσιαστικά μέσω των επαφών αυτών να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση για το τι θα πρέπει να γίνει προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παράνομες αυτές χρηματοοικονομικές ροές και προκειμένου τελικά να εξαλειφθούν. Όπως υπόθηκε και από τους Προέδρους, η έκθεση αυτή υποβλήθηκε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικής τον Ιανουάριο του 2014. 2015 με συγχωρείτε, εγκρίθηκε στη συνέχεια, καθώς επίσης και σχετικές συστάσεις. Επιστρέφουμε λοιπόν σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την σύνοδο εκείνη που έγινε για την Αφρική, η οποία ζήτησε από το πάνελ μας να κάνει κάθε τι το δυνατό προκειμένου να κοινοποιηθούν αυτές οι συστάσεις και να ενθαρρυνθούν ουσιαστικά και οι δικές μας οι χώρες της Αφρικής, καθώς επίσης και στον υπόλοιπο κόσμο, να αρχίσουν τελικά να εφαρμόζουν αυτά τα πορίσματα και αυτές οι συστάσεις. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι συστάσεις αυτές ελήφθηκαν υπόψη και από τη Διεθνή Διάσκεψη Χρηματοδότησης για την Ανάπτυξη τον Ιούλιο του 2015 στην Αντίσα Μπέμπα και στη συνέχεια απασχόλησαν και την σύνοδο του ΟΗΕ του Σεπτεμβρίου του 2015, η οποία ενέκρινε τελικά και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Στα πλαίσια της συνόδου αυτής αναφερθήκαμε και στις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να εξαλειφθούν οι παράνομες αυτές χρηματοοικονομικές ροές. Χαιρόμαστε λοιπόν πολύ ως Ήπειρος πλέον, ως Αφρικανική Ήπειρος που το ζήτημα αυτό απασχολεί το διεθνές προσκήνιο και επιστρέφουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθώντας πλέον να προωθήσουμε έναν στόχο που είναι ένας κοινό πλέον στόχος ανάμεσα σε εμά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν υπό το φως όλων αυτών των αποφάσεων να δούμε ποια θα είναι τα μελλοντικά μας βήματα. θα ήθελα να παραθέσω κάποιες παραγράφους από το έγγραφο συμπερασμάτων της Συνόδου της Αντίς Αμπέμπα, γιατί νομίζω ότι πραγματικά αναφέρονται με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών σε παγκόσμιο επίπεδο. και τι θα πρέπει να γίνει σε σχέση επίσης και με την αναπτυξιακή ατζέντα για την περίοδο μετά το 2015. Πριν από τη Σύνοδο του Σεπτεμβρίου των Ηνωμένων Εθνών. Λέγεται λοιπόν ότι το θεματολόγιο αυτό, το αναπτυξιακό, θα πρέπει να διέπεται από φιλόδοξα και αξιόπιστα μέσα εφαρμογής. είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διατηρήσουμε στην Αφρική όλο αυτό το διαφεύγον κεφάλαιο, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη της Αφρικής. Λέμε λοιπόν ότι από κοινού θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σφαιρικό και διορατικό πλαίσιο, προκειμένου να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε αυτή την αναπτυξιακή ατζέντα, η οποία εμπεριέχει και το στόχο της καταπολέμησης των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Λέμε στη συνέχεια ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε και τη συνένεση του Μοντερέι καθώς επίσης και τη δήλωση της Ντόχα και ότι πρέπει επίσης να ενισχύσουμε το πλαίσιο για την χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς επίσης και να ενισχύσουμε τα μέσα εφαρμογής της παγκόσμιας αναπτυξιακής ατζέντα και ότι θα πρέπει επίσης να αναζωογονήσουμε και να ενισχύσουμε την διαδικασία παρακολούθησης της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη προκειμένου όλες οι δεσμεύσεις μας να εφαρμόζονται στην πράξη και να αξιολογούνται με τρόπο έγκαιρο και διαφανή. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε όντως στους στόχους αυτούς, να επιμείνουμε στο ζήτημα της εφαρμογής των συστάσεών μας. Σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλές ε, συζητήσεις και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη δική μας συμμετοχή για το ότι πραγματικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε εδώ μια πολύ σημαντική πρόκληση, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και ότι πρέπει συνεπώς να έχουμε ένα κοινό υψηλό επίπεδο δέσμευσης προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποφάσεις μας. Και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, η διάσκεψη της Άντις Σαμπέμπα είπε ότι θα πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να μειώσουμε τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές με χρονικό ορίζοντα το 2030 και με απότερο στόχο να τις εξαλείψουμε συμπεριλαμβάνοντα συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τους εθνικούς νόμους, κανόνες, καθώ επίσης και τη διεθνή συνεργασία. Επίσης θα πρέπει να μειώσουμε τις δυνατότητες φόρο αποφυγής και θα πρέπει να δημιουργήσουμε και ρήτρε κατά, κατά των καταχρηστικών πρακτικών σε όλες τις συμφωνίες και τις φορολογικές συμφωνίες και ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις πρακτικές κοινοποίησης δεδομένων και τη διαφάνεια τόσο στις χώρες προέλευση όσο και στι χώρε προορισμού, συμπεριλαμβάνοντα επίση διαφάνεια για όλε τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγές μεταξύ κυβερνήσεων και εταιριών σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία υποβάλλουν στι φορολογικέ αρχέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείε και συγκεκριμένα οι πολυεθνικές εταιρείες καταβάλουν όντως τους φόρους τους στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται και στι χώρε όπου δημιουργούν κέρδο, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνέ δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε επίσης από την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ομένα Έθνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να βοηθήσουν τόσο τις χώρες προέλευσης όσο και τις χώρες προορισμού. Προτάθηκε επίσης στη συνδιάσκεψη αυτή ότι οι περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν εκτιμήσεις όσον αφορά τη σύνθεση αλλά και το μέγεθος των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Οφείλω λοιπόν εδώ πέρα να πω ότι προχθές συζητήσαμε το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα με εκπροσώπους του ΟΣΑ στο Παρίσι και συμφωνήσαμε ότι όντως θα πρέπει να καταφέρουμε να παρακολουθήσουμε περισσότερο τις ροές αυτές, να καταμετρήσουμε τις ροές αυτές, προκειμένου τελικά να είμαστε σε θέση να δούμε αν όντως σημειώνουμε πρόοδο στην ε, καταπολέμηση του φαινομένου αυτού και αν τελικά το φαινόμενο αυτό όντως μειώνεται και αν σιγά σιγά οδεύει προς την ε, τελική του κατάργηση. Αναφερθήκαμε όμως και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό μας απασχόλησε και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πέρυσι. Σε σχέση λοιπόν με το ζήτημα το οποίο συζητάμε εδώ πέρα σήμερα, θα θυμάστε ενδεχομένω μία από τις εκκλήσεις που είχαμε κάνει και είχαμε συμφωνήσει στο παρελθόν, όπου είχαμε πει ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει να μειώσουμε τις ε, παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, καθώς επίσης και τις ε, ροές, ε, παράνομες ροές όπλων και ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή οργανωμένου εγκλήματος. Ένας επίσης σχετικός στόχος έλεγε ότι θα πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν οι εσωτερικοί πόροι μέσω διεθνής υποστήριξης επίσης προς αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να βελτιωθεί και η εγχώρια ικανότητα συλλογής φόρων και άλλων εσόδων. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα σήμερα αξιότιμοι ευρωβουλευτές προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού προκειμένου να καταπολεμήσουμε πλέον ένα φαινόμενο το οποίο είναι παγκόσμιο και προκειμένου να προωθήσουμε έναν στόχο ο οποίο είναι πλέον κοινό καθολικό, η καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Χαίρομαι πάρα πολύ επίση που αναφέρεται και το ζήτημα των ε, εγγράφων του Παναμά, γιατί και στη δική μα την έκθεση, όπω θα το έχετε άλλωστε δει, αναφερόμαστε στο ζήτημα αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι πάρα πολλέ από τι παράνομε αυτέ χρηματοοικονομικέ ροέ απορρέουν τελικά από φορολογικού παραδείσου ή από δικαιοδοσίε οι οποίε παρέχουν δυνατότητε χρηματοοικονομικού απορρίτου. Ακριβώ λοιπόν αυτό πρέπει να μα απασχολήσει. Τι μπορούμε εμεί να κάνουμε προκειμένου να εξαλείψουμε τις πρακτικές αυτές διατήρηση εσόδων, προσόδων, πιο συγκεκριμένα σε φορολογικούς παραδείσους και σε δικαιοδοσίε που παρέχουν χρηματοοικονομικό απόρριτο. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το γεγονό ότι δεν υπάρχει διαφάνεια ω προ το ποιο είναι ο πραγματικό δικαιούχο διαφόρων επιχειρήσεων. Και οι πληροφορίε οι οποίε απορρέουν πλέον από τα έγγραφα του Παναμά ουσιαστικά επιβεβαιώνει και τα δικά μα τα πορίσματα, αυτά τα οποία μπορείτε να δείτε στην έκθεσή μα, ότι όντω πρέπει να βάλουμε κατά του δικτύου αυτού υπεράκτιων λογαριασμών και ότι θα πρέπει να αποθαρρύνουμε οποιαδήποτε παράνομη τέτοια μετακίνηση εσόδων προς φορολογικούς παραδείσους. Το ζήτημα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βαθύνει περισσότερο στο ζήτημα αυτό των φορολογικών παραδείσων και των δικαιοδοσιών που παρέχουν, που προσφέρουν χρηματοπιστωτικό απόρριτο και τι μπορεί να γίνει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να παταχθούν τα φαινόμενα αυτά. Και επίσης να δούμε τι μπορεί να γίνει και με το ζήτημα του πραγματικού δικαιούχου. Να μπορούμε να βλέπουμε δηλαδή ποιος πραγματικά υποφελείται από την επιχειρηματική δραστηριότητα συγκεκριμένων εταιριών. Ως προς αυτό, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε Καταρχά, ποιο είναι ο πραγματικό δικαιούχο, ποιο πραγματικά ωφελείται από τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, αλλά πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένα δημόσια και διαφανή μητρώα για αυτέ τι επιχειρήσει. Πριν από δύο χρόνια περίπου, ζητήσατε από την υψηλόβαθμη ομάδα μας να έρθουμε σε επαφή με αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό του beneficial ownership, του πραγματικού δικαιούχου. Το πράξαμε αυτό. Λάβαμε λοιπόν κάποιες απαντήσεις, ορισμένες από τις οποίες ήταν ότι ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να ασχοληθούμε με το ζήτημα του πραγματικού δικαιούχου, ωστόσο μας λέγανε ότι όσον αφορά το ζήτημα των ε, ταμείων δεν μπορούμε να τα περάσουμε σε ένα δημόσιο μητρό. Αυτό μας είπανε και χρησιμοποίησαν ένα επιχείρημα το οποίο δεν καταλάβαμε πολύ καλά. Ευτυχώ όμως βλέπω ότι ακόμα και για το ζήτημα αυτό υπάρχει μια αλλαγή κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και για τον πραγματικό δικαιούχο όμω των επιχειρήσεων, γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αναλάβουμε τη δέουσα δράση. Είμαστε λοιπόν πεπισμένοι ότι η δημοσιοποίηση των εγγράφων του Παναμά, αν μη τι άλλο, είχε το εξή θετικό ότι αυξήθηκε η ευαισθητοποίηση και η γενικότερη γνώση πλέον που υπάρχει παγκοσμίω όσον αφορά την ευρύτερη αυτή χρησιμοποίηση φορολογικών παραδείσων και δικαιοδοσιών που παρέχουν χρηματοπιστωτικό απόρριτο, προκειμένου να διαφύγουν πόροι και κεφάλαια τα οποία θα έπρεπε λογικά, όπως είπε και η Συμπρόεδρος, να ήταν ε, διαθέσιμα στις αναπτυσσόμενες χώρες για την ε, δική τους εγχώρια ανάπτυξη. Και αν ήταν διαθέσιμη όντως οι πόροι αυτοί και μέναν σε εθνικό επίπεδο, δεν θα αναγκάζονταν τόσοι πολλοί άνθρωποι να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό και να εγκαταλείψουν την Αφρικανική Ήπειρο. Θα ήθελα να χαιρετήσω την πολύ σημαντική εργασία που έχει γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το ζήτημα της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Θεωρούμε ότι οι πρωτοβουλίες αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Ελπίζω ότι ε, θα ευοδοθεί η πρωτοβουλία αυτή και παράλληλα θα πρέπει να δούμε βέβαια ποια είναι η διοικητική ικανότητα των ίδιων των Αφρικανικών κρατών να χρησιμοποιήσουν αυτό το αυτόματο σύστημα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνατότητες συλλογής φόρων. Τώρα το ζήτημα της εφαρμογής της υποβολής εκθέσεων αναχώρα, country by country reporting. Και αυτό το ζήτημα έχει απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είπατε ότι η υποβολή αυτή εκθέσεων αναχώρα θα πρέπει να ισχύει και για τις εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και αν δεν κάνω λάθος, η υποχρέωση αυτή ήδη υφίσταται για τις τράπεζες και αυτή τη στιγμή εξολογείται όταν θα πρέπει επίση να ισχύει και για τι πολυεθνικέ επιχειρήσει. Το σύστημα αυτό υποβολή εκθέσεων να χώρα αποτελεί πολύ σημαντικό μέρο του συστήματο καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Γνωρίζετε πολύ καλά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μη διαφοροποιημένες μεθόδου δημοσιοποίηση των εσόδων το επιτρέπουν τελικά σε πάρα πολλές επιχειρήσεις να αποκρύβουν μέρος των εσόδων τους. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εργασία που έχει κάνει σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Σαφώς πιστεύω ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ιδίως εμείς στην Αφρικανική Ήπειρο, είναι το ζήτημα της αδυναμίας των θεσμών μας και της έλλειψης διοικητικών ικανοτήτων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Θα θέλαμε λοιπόν ως προς αυτό να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η συνεργασία αυτή έχει να κάνει ουσιαστικά με ζητήματα που είναι πλέον νομοθετικά, γιατί πέρα από τα ίδια τα θεσμικά όργανα και πέρα από του διοικητικού υπαλλήλου που θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, χρειαζόμαστε και το απαραίτητο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να μπορέσουμε αποτελεσματικά να καταπολεμήσουμε τι παράνομε αυτέ χρηματοοικονομικές ροέ. Η εμπειρία λοιπόν που έχει συσσωρεύσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το νομοθετικό του έργο για τον κλάδο αυτό, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και τι αφρικανικέ χώρε προκειμένου να καταφέρουν να ενισχύσουν τη διοικητική του ικανότητα. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι ε, το ζήτημα της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας, ακόμα και σε σχέση με τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια νομοθεσία ή την περαιτέρω βελτίωσή τους, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε δηλαδή ποια είναι τα συγκεκριμένα συμπεράσματα στα οποία έχετε καταλήξει εσείς, ποια είναι τα ωφέλη και ποιες είναι οι προκλήσεις από την υιοθέτηση μιας τέτοιας νομοθεσίας. Η συνεργασία μας λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ζητήματα αυτά, αυτή η ανταλλαγή εμπειριών θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή διοικητική ικανότητα για τις χώρες της Αφρικής προκειμένου να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο η δράση μας θα είναι πραγματικά αποτελεσματική και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να μειώσουμε και να εξαλείψουμε εν τέλει το φαινόμενο αυτό των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Από αφρικανικής λοιπόν σκοπιάς δεν μπορούμε πλέον να λέμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι καθαρά αφρικανικό. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι επιτρέπουμε εμείς σε πάρα πολλά κεφάλαια να διαφεύγουν από την Αφρικανική Ήπειρο, επομένω πρέπει σε αφρικανικό επίπεδο να λάβουμε δράση εμείς, αλλά σίγουρα πρέπει να παραδεχθούμε παράλληλα ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο πλέον. Ως προς αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η θεσμική συνεργασία μεταξύ ημών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χάρηκα πάρα πολύ όταν οι συμπρόεδροι αναφέρθηκαν στην έκθεση την οποία υποβάλαμε και είδα και έναν ευρωβουλευτή ο οποίος μπήκε στην αίθουσα κρατώντας το έγγραφο αυτό. Αυτό με χαροποίησε όλος ιδιαιτέρως. Σας καλώ λοιπόν, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μελετήσετε πραγματικά αυτή την έκθεση. Να δείτε όλες τις συστάσεις, όλα τα πορίσματα της έκθεσης αυτής, αφενός με ένα. Διότι ε, η διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης πέρασε πάρα πολύ χρόνο ασχολούμενη με το ζήτημα αυτό και τελικά κάλυψε τα ίδια ζητήματα με εμάς. Και αφετέρου γιατί γίνονται και κάποιες πάρα πολύ σωστές προτάσεις για το, για το τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, που συνδέεται, όπως σας είπα, και με την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, χρειάζεται μια παγκόσμια δέσμευση για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Πήγαμε λοιπόν και στην Ουάσιγκτον, συνομιλήσαμε με εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συζητήσαμε και με εκπροσώπους της Αμερικανικής Κυβέρνησης, με εκπροσώπους της ΕΚΟΣΟΚ των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη Άλλωστε γνωρίζετε ότι είναι αυτοί οι πλέον αρμόδιοι για να δούνε πώς θα εφαρμόζονται τα μέτρα μας για το ζήτημα αυτό, τα μέτρα καταπολέμησης δηλαδή των χρηματοοικονομικών ροών. Προχθές, όπως σας είπα, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους του ΟΣΑ στο Παρίσι. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω ότι θα έχουμε συνομιλίες και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αύριο μάλιστα θα συναντηθούμε με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φραγκφούρτη. Στόχος όλων αυτών των επαφών είναι να κινητοποιηθούμε όλοι προκειμένου να λάβουμε δράση κατά του φαινομένου αυτού. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε κανένα κενό ή καμία έλλειψη στη δράση μας. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συντονισμένοι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο γιατί μόνο η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού θα οδηγήσει στην ίσπραξη όλων αυτών των εσόδων που πρέπει ουσιαστικά να έχει Αφρικανική Ήπειρος. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει να διατηρήσει σε χώριο επίπεδο τους πόρους της που θα χρησιμοποιηθούν για την εσωτερική ανάπτυξη της Αφρικανικής Ήπειρου και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε χιλιάδες άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο προσπαθώντας να εγκατασταθούν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να ανταλλάξω απόψει μαζί σα να δω ποια είναι η δική σα η άποψη σε σχέση με τα μέτρα τα οποία πρέπει να υιοθετήσουμε για να πατάξουμε το φαινόμενο των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Βλέπετε ότι το ζήτημα αυτό πλέον δεν είναι μόνο περιφερειακό, αλλά απασχολεί την παγκόσμια οικονομική και αναπτυξιακή ατζέντα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα η πρόεδρος κυρία Μακάβαν. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση του θέματος που μας προσφέρει τροφή για σκέψη πράγματι. Χρειάζεται να δώσουμε συνέχεια στην εργασία μας. Και βέβαια στους ε, θεσμικούς συνδέσμους θα το εξετάσει η Επιτροπή μας πώς μπορούμε να το προωθήσουμε διότι ορισμένοι που παρακολουθούν θα πούν «Α, ωραία λόγια, τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα» αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε βέβαια είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Να πείσουμε τις κυβερνήσεις ότι τώρα κάτι πάει να γίνει και χρειάζεται ένα συγκεκριμένο follow-up. Έχουμε και την Επιτροπή μας, έχουμε και την Επιτροπή Εξωτερικών αλλά και την Επιτροπή Οικονομικών που όλοι αυτοί εξετάζουν το θέμα των παράνομων χρηματικών εργών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να ανακοινώσει νέα μέτρα. Έχουμε αρχίσει τώρα την ε, διαδικασία, προάγουμε τη διαδικασία για την ε, υποβολή εκθέσεων αναχώρα, αλλά μόνο για ε, τα ορυκτά. Να επεκταθεί λοιπόν. Υπάρχει τώρα το παράθυρο ευκαιρίας και αυτό ε, είναι που πρέπει να δούμε με πιο συγκεκριμένο τρόπο δηλαδή θα προχωρήσουμε. Θα αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση. Θα δώσω πρώτα τον λόγο στη συνάδελφό μου Σλάιν που έχει κάνει και τη σχετική έκθεση. Έλλη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μπέκε για την πολύ σημαντική τοποθέτησή σας. Όπως είπατε, με το σκάνδαλο των εγγράφων του Παναμά κατέστησα φες ότι είναι παγκόσμιες πλέον οι διαστάσεις ε, της πρόκλησης. Δηλαδή με μονομένες χώρες μέλη της Ένωσης ή άλλες χώρες εταίροι ούτε καν διανοούνται ότι μπορούν να το αντιμετωπίσουν μόνες τους όπως Σέρα Λεόνε, Ουγγάντα, Νότια Αφρική, ε, Νιγηρία είναι κάποιες από τις χώρες που αναφέρονται μέσα στην ε, έρευνα για την για την οργάνωση ΦΟΝΣΕΚΑ που έχει, ε, βρίσκεται δηλαδή στην αρχή αυτή τη ιστορία των εγγράφων του Παναμά. Οι προκλήσει είναι τεράστιε, το είπε και ο κύριο Μπροκ. Και αυτό, είναι, αυτό σημαίνει ότι και εμεί να κάνουμε τεράστιε προσπάθειες για να διευκολύνουμε την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στι χώρε αυτέ. Πέρσι, ω εισηγήτρια, για την έκθεση σχετικά με τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή στι αναπτυσσόμενε χώρε. δουλέψαμε πολύ πάνω στο θέμα αυτό, οι προκλήσεις ό,τι αφορά την διαχείριση, ε, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη. Εγκρίθηκε πριν από την διάσκεψη για την ε, οικονομική ανάπτυξη. Όμως, εξακολουθεί το βασικό πρόβλημα να είναι ότι οι εγχώροι πόροι θα είναι πάντα η βασική πηγή χρηματοδότησης των χωρών αυτών. Και αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ε, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή θα έχουμε υψηλέ αποδόσεις από την ίσπραξη των φόρων και ενίσχυση επομένω των θεσμών και των ε, κυβερνήσεων. Στην έκθεσή μου ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες τον αγώνα τους αυτό, προσφέροντας οικονομική και τεχνική βοήθεια, διότι η βοήθεια για τα θέματα αυτά εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, κάτω από το 1% το 2011. Σε ό,τι αφορά τη συνολική βοήθεια. Έγιναν κάποια βήματα στην Άντις Αμπέμπα. Είδαμε και τη σχετική πρωτοβουλία για τα φορολογικά. Ε, υπάρχει πρόβλημα και με τις ε, συνθήκες δημοσιονομικού χαρακτήρα διότι δεν γίνονται πάντα σωστά οι κατανομές των εσόδων μεταξύ χωρών υποδοχής και χωρών προέλευσης. 500 από αυτές τις ε, συνθήκες εξετάστηκαν. Εμείς προτιμούμε βέβαια τη συνθήκη που βασίζεται στα πρότυπα, δηλαδή τα πρότυπα μάλλον, των Ηνωμένων Εθνών και όχι του ΩΣΑ. Ε, ζητούσαμε επίσης να γίνονται μελέτες αντικτύπου αυτό ορισμένες χώρες το κάνουν ήδη, όπως η Ολλανδία, που να δείχνουν ποιες είναι οι επιπτώσεις των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών πολιτικών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη, της Ολλανδία δείξανε ότι υπάρχουν επιπτώσεις της τάξης των 500 έως 700 εκατομμυρίων το χρόνο. Τώρα, ακόμα και αν υποστηρίξουμε τις προσπάθειες του ΟΟΣΑ και όλη την διαδικασία που ονομάζεται BEPS, δηλαδή διάβρωση φορολογικής βάσης και μετακίνηση κέρδων, σημαίνει πάντως πολύ, ανάγκη μάλλον πολύ μεγαλύτερης συμμετοχής των αναπτυγμένων χωρών. Αυτό ζητούσαμε πάλι στην εκθεσή μου. Και τέλος, ως ένα βασικό εργαλείο για τη διαφάνεια, πολύ σωστά είπατε και εσείς, στοχεύσαμε στην ανάγκη απόλυτης διαφάνειας ό,τι αφορά τους πραγματικούς ιδιοκτήτε, πραγματικού δικαιούχου των διαφορών επιχειρήσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι κρίσιμη σημασία μεν. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε ωστόσο αμοιβαιότητα διότι οι ορισμένε χώρε σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα να ε, κάνουν την ανταλλαγή των πληροφοριών με τον ίδιο τρόπο που σε ευρωπαϊκέ χώρε. Χρειάζεται λοιπόν μια μεταβατική περίοδο μέχρι να φτάσουμε σε πλήρη λειτουργία τη ε, αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Και τέλο, ένα δημόσιο σύστημα υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάποια βήματα προς τα εμπρός για να διασφαλίσει την διαφάνεια. Ωστόσο, χάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια σημαντική ευκαιρία και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας εκεί, διότι η πρόταση για το CBCR έχει όρια, όρια μάλιστα αυστηρά. Δεν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια για το τι πράττουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Επικράτειας των Ευρωπαϊκών χωρών μελών. Γνωρίζουμε επίσης ότι θα είναι συνολικά δεδομένα, τα οποία ασφαλώς και δεν αρκούν. Τέλος, το κατόφλι των 750 εκατομμυρίων κύκλου εργασιών της επιχειρήσεως, από το οποίο και μετά υποχρεούται να υποβάλει τις εκθέσεις στη βάση του συστήματος που προβλέπεται. Εμείς θεωρούμε ότι το κατόφλι αυτό είναι υπερβολικά υψηλό. Άρα υπάρχουν όρια σε αυτό το σύστημα ε, CBCR. Πρέπει να κάνουμε σημαντικές προσπάθειες για να στηθεί στα πόδια του ένα σύστημα το οποίο να αντιμετωπίζει τις ανάγκες αυτές και μάλιστα σύντομα. Όπως είπαν και άλλοι συναδελφοί μου, όταν μιλούμε για συνοχή πολιτικών ανάπτυξης, βέβαια θέλουμε να χτυπήσουμε, μάλλον θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τη ρίζα και των μεταναστευτικών ροών για να αντιμετωπίσουμε βέβαια όλες αυτές τις δυσκολίες που βλέπουμε καθημερινά. Σημειώστε εγώ είμαι Ιταλίδα. Δεν αρκεί να εργαστούμε πάνω σε μεταναστευτικές πολιτικές, πρέπει να εργαστούμε περισσότερο και καλύτερα και πάνω σε πολιτικές ανάπτυξης αλλά και σε δημοσιονομικές πολιτικές που είναι προφανές ότι έχουν επιπτώσει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Έλλη για την ενημέρωση για το τι συμβαίνει εδώ. Και τώρα ο κύριος Στίερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο Εμπέκε για την ε, τοποθέτησή του και τον ευχαριστώ που έχει προσέλθει εδώ ενώπιόν μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα συνεχίσω λίγο πολύ πάνω στην γραμμή της ε, Ellis Line. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι μόνο ε, δημοσιονομικού χαρακτήρα, ούτε μόνο αναπτυξιακού, ούτε μόνο οικονομικού χαρακτήρα. Είναι όλα αυτά, αλλά κυρίως είναι πολιτικό πρόβλημα. Και επομένως απαιτεί πολιτική λύση. Η έκθεσή σας επιβεβαιώνει άλλωστε ότι τα ποσά των παράνομων χρηματικών ροών είναι περίπου δεκαπλάσια από την επίσημη ε, οικονομική βοήθεια. Για κάθε ευρώ που φέρει από την Ευρώπη για να πάει στην Αφρική ως βοήθεια, 10 ευρώ φεύγουν παράνομα από την Αφρική. Δεν μιλούμε μονάχα για ε, παράνομες ροές εξόδου, είναι παράνομος και ο τρόπος με τον οποίο παρήχθη το χρήμα αυτό. Όταν μιλούμε λοιπόν για παράνομες χρηματικές ροές, μιλούμε εν τέλει για διαφθορά. Και όταν μιλούμε για διαφθορά, είπατε σωστά κι εσείς, ότι χρειαζόμαστε κάποιες παγκόσμιες λύσεις όπως ε, country by country reporting και άλλα κάποια στοιχεία, τα αναφέρατε κι εσείς, αλλά είπατε κάτι άλλο ακόμη που είναι σημαντικό είναι δηλαδή η αδυναμία των κρατικών θεσμών, η έλλειψη συμπερίληψης και στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο, διότι η έλλειψη συμπερίληψης, inclusiveness δηλαδή, προωθεί και τη διαφθορά. Και αυτό είναι διότι υπάρχει μια πολιτική επικυριαρχία, ένα πολιτικό πατρονάρισμα, το οποίο επιτρέπουν οι θεσμοί. Δεν υπάρχει δηλαδή χρηστή δημοκρατική διοίκηση και διαχείριση. Βλέπουμε πολιτικές δυνάμεις οι οποίες είναι κατεστημένες στην εξουσία παραπάνω από 20 χρόνια σε διάφορες χώρες, σε ορισμένες αφρικανικές χώρες, χωρίς να γίνεται καμιά αλλαγή. Και αυτό βέβαια προκαλεί την διαφθορά. Το ερώτημα λοιπόν για μας όλες και όλους εδώ είναι συζητούμε τώρα για παράδειγμα τι θα κάνουμε μετά την εκπνοή της ε, Συμφωνίας Κοτονού, τι θα κάνουμε δηλαδή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων μας, των χωρών ΑΚΕ. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε το επόμενο βήμα για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού και βέβαια και της πολιτικής του διάστασης, της ε, ορθής πολιτικής διακυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν τελικά οι παράνομε χρηματικές ροές και ποια θα είναι τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτό. Μπορούμε να επιμείνουμε σε μια διαρθρωμένη εφαρμογή της αρχής more for more, δηλαδή περισσότερα έναντι περισσότερων στη συνεργασία μας και για θέματα βέβαια αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτά θα μπουν στον πυρήνα της συζήτησης. Επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό έχει ένα έντονο πολιτικό χαρακτήρα και χρειάζεται πολιτικές λύσεις. Ευχαριστώ, κύριε Γκόμες. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Είμαι μέλος της Επιτροπής μας που την έχουμε αποκαλέσει ΤΑΞ 2 και είχε αρχίσει, ε, είχε δημιουργηθεί μάλλον με την ε, αφορμή του προηγούμενου σκανδάλου των διαρροών του Λουξεμβούργου πριν από τον, τις του Παναμά. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε. Όπως είπατε άλλωστε υπάρχει περιορισμένη συνάρθρωση μεταξύ μας. Μπαίνουμε τώρα, έχουμε και άλλη δηλαδή επιτροπή ε, με ε, αρμοδιότητες Εξεταστικής Επιτροπής για τα έγγραφα του Παναμά. Εγώ θα ήθελα να δω πολύ περισσότερες επαφές μαζί μας. Ιδίω, εσείς περιγράψατε και αναλύσατε το πρόβλημα. Εμείς αναλύσαμε επίσης το πρόβλημα στην πρώτη μας έκθεση της πρώτης Επιτροπής Τάξης και το αναλύουμε πάλι στην έκθεση της δεύτερης Επιτροπής Τάξης. Γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει. Ε, γνωρίζουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για συγκεκριμένες υποθέσεις όπου πρέπει να επιφέρουμε κάποια διαφορά. Και εκεί αυτό θα απαιτήσει και τη συνεργασία σας. Και μάλιστα να εργαστούμε ταχαίως, διότι όπως είπαν οι δύο προηγούμενοι συνάδελφοι, το πρόβλημα είναι πολιτικό. Και υπάρχει πάρα πολύ συνάρθρωση, διασύνδεση μεταξύ της δικής σας διαφθοράς και της δικής μας διαφθοράς. Εδώ το σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι, ώστε να προκαλεί διαφθορά. και τρέφει όλη αυτή την βιομηχανία συμβούλων, ε, νομικών συμβούλων, δικηγόρων και ούτω καθεξής για, ε, και φτάνει και απολύγει σε όλες αυτές τις ε, περίφημες ε, ε υπεράκτητες εταιρείε. Πρόκειται εν τέλει για οργανωμένο έγκλημα και σε αυτό εντάσσω και την τρομοκρατία. Ο αγώνας μας λοιπόν υπέρ της ακαιρεότητας συνεπιφέρει, συνεπάγεται και τον αγώνα κατά τη τρομοκρατία, που είναι ζήτημα επιβίωση για τι κοινωνίε μα και βεβαίω για τι κυβερνήσει και στην Αφρική όπω και στην Ευρώπη. Η δε πρόφαση ότι, α, κοιτάξτε, αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο στο παγκόσμιο επίπεδο, ε, αυτά δεν τα δέχονται πλέον οι πολίτε μα. Θα πρέπει βεβαίω να κάνουμε ό,τι μπορούμε εμεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στην Αφρική μαζί σα, αλλά πρέπει να δούμε και τους συναδελφούς μας των Ενωμένων Πολιτειών. Ας αρχίσουμε όμως κάπου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ερωτήσω πέραν αυτών ω εξή. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένε υποθέσει. Εγώ εργάζομαι επί συγκεκριμένων υποθέσεων εκεί, όπου η χώρα μου, η Πορτογαλία, λειτουργεί ω πλυντήριο για χρήματα που έρχονται από την Αγγόλα, για παράδειγμα, και από άλλε χώρε τη Αφρική, Νιγηρία και αλλού, το Βέλγιο, ενδεχομένα για την λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και αλλού. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Ρωτώ λοιπόν, τι θα κάνουμε για να προστατεύσουμε τους καταγγέλλοντες, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, διότι αυτά τα πρόσωπα βρίσκονται στην απαρχή των καταγγελιών, ανοίγουν τα μάτια των πολιτών μας και στην Ευρώπη όπως και στην Αφρική. Τι κάνουμε λοιπόν για να προστατεύσουμε αυτούς που στα αγγλικά τους λένε whistleblowers διότι αλλιώ, αν δεν κάνουμε τίποτα, καταδικάζονται σε σιγή. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος Μακάβαρα, ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ επίκαιρη η επίσκεψή σας, το είπαν και πολλοί από τους προλαλήσαντε συναδέλφους και νομίζω ότι πολύ σωστά επισημάνατε το γεγονός ότι θα πρέπει ε, να επιτελείτε το έργο και στις χώρες ε, προέλευσης και στις χώρες προορισμού. Και είδατε κι εσείς ε, ότι γίνονται πολλά αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε και τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκθέσεις αναχώρα. Είμαι βέβαιο ότι το Κοινοβούλιο θα βελτιώσει αυτή την πρόταση που είναι καλή αρχή μεν, αλλά δέχεται βελτιώσει. Το είπε και η Έλλη Σλάιν. Αυτό που θέλω να πω, ε, νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτό που είπε ο συνάδελφος Στυρ. Δηλαδή, ήρθε η ώρα πλέον να, να ε, τονίσουμε τη σημασία της ε, καλής διακυβέρνησης και της λογοδοσίας στις χώρες προέλευσης. Έχω μια ερώτηση. Εάν κάποιες από τις εθελοντικές πρωτοβουλίες, η ITI για παράδειγμα, μπορούν αυτές να επεκταθούν και να, κατα... Ε, να αναφέρονται και στους φυσικούς πόρους, τα δάση για παράδειγμα, διότι νομίζω ότι και τα δάση είναι αντικείμενο πολλών ε, παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και πολλής διαφθοράς. Δεν ήταν καλό ή εν λόγω πρωτοβουλία κάποια νέα πρωτοβουλία να αναλυφθεί για τα δάση στην Αφρική. Δεύτερη ερώτηση, να συμφωνήσω και με την ε, ανάλυση πάλι του κυρίου Στίαρ, ότι βλέπουμε κυβερνήσεις, προέδρους ε, που ε, ήταν 20 χρόνια πρόεδροι και σχεδιάζουν να παραμείνουν στην εξήγη ακόμα 20 χρόνια. Βλέπουμε ότι πολλές φορές με την ισχυρή αυτή προεδρική ηγεσία έχουμε κρατική ε, ιδιοκτησία και πολλές χρηματοοικονομικές ροές εκεί κάπου ε, εντοπίζονται, όπως ε, με τη, δημοκρατική, τη λαϊκή συγγνώμη, δημοκρατία του Κονγκό, που ο πρόεδρος νομίζω είχε κάποιες επαφές με κάποια εταιρεία μεταλλευμάτων από, τη, από το Καζακστάν που είχε έντρα στο Λονδίνο, μια άλλη, ένας Ισραηλινός επιχειρηματίας που μεσολαβούσε κτλ. Και νομίζω ότι ε, το ποσό αντιστοιχούσε στο διπλάσιο του εκπαιδευτικού προϋπολογισμού της χώρας. Επίσης, πριν από δύο χρόνια στο Financial Times λέγεται ότι ένα ε, δις ε, ευρώ διεθνών δανείων είναι ένα ποσό, παραδείγματος χάρη εταιρείε που υποτίθεται ότι αλλιεύουν τόνο κτλ. Αλλά τελικά προστατεύουν τις τεράστιες επιχειρήσεις εξόριξη πετρελαίου εκτός Μοζαμβίκης και υπάρχει μια πραγματική κρίση στη χώρα. Πιστεύετε ότι έχουμε και στην περίπτωση αυτή παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Τέτοια συμβάντα πραγματικά αμφισβητούν και την ολεξοπιστία μιας κυβέρνησης. Ευχαριστώ, Ιγνάσιο Κοράου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο Μπέκη για την παρουσία του σήμερα στις επιτροπές μας. Σύμφωνο με τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και φυσικά μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ένα πολιτικό πρόβλημα για το οποίο βέβαια απαιτούνται παγκόσμιες και πολιτικές λύσεις. Όταν ε, μιλούμε για παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, δεν μιλούμε μόνο για την Αφρική. Φυσικά είναι μεγάλες οι απώλειες ε, στην Αφρική, γιατί θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η φτώχεια με αυτά τα χρήματα. Αλλά μιλάμε για απώλειες και στον κόσμο τον υπόλοιπο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ άλλων και συμφωνώ με την ανάλυση της συναδέλφου Άννα Γκόμες, η οποία είπε ότι ε, σχετίζεται το όλο θέμα με τη διαφθορά. Και εγώ θα έλεγα ότι σχετίζεται και με το οικονομικό μοντέλο, όπου βλέπουμε ε, τα κεφάλαια να ε, κατευθύνουν και να ορίζουν την πολιτική. Επειδή συζητούμε για την Αφρική, ε, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές το 2000 στο 2010 ήταν πετρέλαιο, μεταλλεύματα, χαλκός, χάλιβας, σίδηρος και ε, υπάρχει σίγουρα δικαιοδοσία, υπάρχουν δικαιοδοσίες που παρέχουν χρηματοπιστωτικό απόρριτο και έχουμε και δραστηριότητες ξεπλήματος χρήματος. Ε, είναι καταστροφικές συνέπειες όλων αυτών και υπάρχουν ε, σημαντικές επιπτώσεις. Τις βλέπουμε και στην κοινωνική πραγματικότητα, δύο τεράστια κεφάλαια απορροφώνται, ενώ αυτοί οι πόροι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον αγώνα κατά της φτώχειας και να τονώσουν την ανάπτυξη των χωρών. Είναι γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη ε, δεν επιθυμούν, νομίζω, πραγματικά να αλλάξουν, να αλλάξουν την πραγματικότητα αυτή ή τέλο πάντων δεν έχουν δείξει τόσο μεγάλη προθυμία. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε όλες οι πολυεθνικές εταιρείες να αποκαλύπτουν δημοσία τα έσοδά τους, τις απώλειες, τα κέρδη, ε, τις επιδοτήσεις ε, και ε, τα επίπεδα του προσωπικού στο πλαίσιο εκθέσεων αναχώρα και να αποφεύγονται πρακτικές, καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές. Επίσης, όλες οι χώρες θα πρέπει να συμμετέχουν στην παγκόσμια προσπάθεια αυτόμας ανταλλαγής ε, χρηματοοικονομικών πληροφοριών για να μην γίνονται μεγαλύτερες καταχρήσεις, εμπορικές συναλλαγές με πολιτικούς παραδείσους και τέτοιες ε, δικαιοδοσίες. Εκεί θα πρέπει να έχουμε το μέγιστο δυνατό ε, επίπεδο ελέγχου από τους φορολογικές και κρατικές αρχές. Θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια. Θα πρέπει να βλέπω το πραγματικό ιδιοκτήτη και δικαιούχο των εταιριών εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη-μέλη που συνεισφέρουν στην περίπτωση φοροδιαφυγής, εξεπλήματος χρήματος, σηματοδότη τρομοκρατίας, ανάπτυξη παραστατιωτικών δυνάμεων και βοήθεια επιδοτής προς ιδιωτικές εταιρείες. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο διαφανές σύστημα, στο οποίο η τίνη επενδυτέ και επιχειρηματίες θα μπορούν να αναπτύσσουν ε, με μεγαλύτερη ασφάλεια τι δραστηριότητε του. Όλε οι πολυεθνικέ, όπω ε, λέγει για παράδειγμα, θα πρέπει να δημοσιεύουν το ισολογισμού, κέρδη από όλε και τα λοιπά, ε, φόρους όπου αναπτύσσουν τη δραστηριότητά του. Αυτό θα διευκολύνει τη δουλειά των αρχών που προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Thanks very much. And uh, our last question is... Τελευταία, η κυρία Χόιμπουρ. Μαρία, παρακαλώ. Μέχρι στιγμής μόνο αγγλικά έχουν ακούσει, αλλά έχουμε Κροάτες, Ιταλούς, Πορτογάλους, συναδέλφους. Ε, ε, όλοι έχουν μιλήσει μέχρι τώρα και από τη Φιλανδία. Συνάδελφος μίλησε. Εσείς θα μιλήσετε γερμανικά. Ναι, θα μιλήσω γερμανικά γιατί είναι και πιο εύκολο για μένα, και χόιμπου. Ε, θα μιλήσω γερμανικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Πρόεδρε Εμπέκη, που έχετε έρθει εδώ ενώπιόν μας. Μιλήσαμε για διαφθορά, για παράνομες ε, οικονομικές δραστηριότητες, για την ανάγκη διαφάνειας. Είπε η Σλάιν, δεν ξέρουμε τι κάνουν οι πολυεθνικοί όμιλοι εκτός Ευρώπης, αλλά δεν ξέρουμε και όλα θα κάνουν εντός Ευρώπης, προσθέτω εγώ. Ήθελα λοιπόν όμως να τονίσω ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν ακούστηκε ως τώρα. Έχουμε πολλές συμφωνίες οικονομικού χαρακτήρα, βεβαίως και με την Αφρική, και σε αυτές τις συμφωνίες η προσπάθεια που γίνεται είναι να δημιουργείται ένα κλίμα θετικό για τις μεγάλες επενδύσεις που θα έλθουν από έξω από την Αφρική. Νομίζω ότι δεν είναι αρκετά δεσμευτικές ωστόσο οι διατάξεις σχετικά με την συμπεριφορά των επενδυτών αυτών και σε ό,τι αφορά δηλαδή την πληρωμή φόρων αλλά και τον σεβασμό τους σε κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά πρότυπα. Εάν δεν περιλάβουμε τέτοιες διατάξεις στις συμφωνίες αυτές, αυτό νομίζω ανοίγει περιθώρια για παράνομες δραστηριότητες. Καμιά φορά μάλιστα και νόμιμες μεν δραστηριότητες που δεν προσφέρουν όμως κανένα πλεονέκτημα στους ντόπιου. Οι οικονομικές αυτές συμφωνίες αποτελούν εν πάση περιπτώσει την βάση για μια κοινή οικονομική διεθνή δράση. Η ερώτησή μου έχει ως εξής. Δεν είναι δυνατόν να κάνετε μια προσπάθεια και σε αυτό το επίπεδο ε, να βάλετε περισσότερο μέσα ε, ε, μια διάσταση δεσμευτικότητας. Και όπως είπε και ο προηγούμενος συναδελφός μου, Κοράου, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες τους οποίους θα οφείλουν να τηρούν οι επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος Μακ Άβαν ε, πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, κύριε Εμπέκη, και για τη συνεργασία και το καθεξής. Κύριε Εμπέκη, έχετε το λόγο. Άκουσα λοιπόν τις ερωτήσεις σας. Ίσως θα πρέπει καταρχάς να πω, κυρία Πρόεδρε, Ως ομάδα υψηλού επίπεδου μας ζητήθηκε από την Αφρικανική Ένωση και συγκεκριμένα από τους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης να υποβάλουμε τις εκθέσεις. Ετήσεις λοιπόν εκθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή από τις αφρικανικές χώρες των όσων συμφωνήθηκαν. Το αναφέρω αυτό διότι στην πράξη αυτό σημαίνει ότι καθήκον μας είναι να πούμε ότι στη χή χώρα, για παράδειγμα, υφίσταται η κατάλληλη νομοθεσία προκειμένου να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Υφίστανται οι κατάλληλοι θεσμοί στη χώρα αυτή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο το οποίο συζητάμε σήμερα. Ο κύριος Στίερ αναφέρθηκε σε αυτό και εφόσον υπάρχουν οι θεσμοί αυτοί είναι επαρκώς διαφανείς, λογοδοτούν επαρκώς, είναι αποτελεσματικοί. Μήπως είναι και οι ίδιοι μέσω περαιτέρω διαφθοράς, μήπως ευνοούν ή διευκολύνουν τη διαφθορά. Αναφέρομαι στα θεσμικά όργανα των κρατών. Είναι λοιπόν σαφές και αυτό άλλωστε λέμε και εμείς στην έκθεσή μας, εργαζόμενοι με τις αφρικανικές χώρες, ότι πρέπει όλο το φάσμα των κρατικών αρχών να είναι συντονισμένο. Αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Τράπεζα, στις φορολογικές αρχές, στις αστυνομικέ δυνάμεις, στις διοκτικές αρχές, και χρειάζεται λοιπόν η απαραίτητη συνεργασία ανάμεσα σε όλε αυτέ τι αρχέ, γιατί σε ορισμένε περιπτώσει μπορεί να υφίστανται τα θεσμικά όργανα, αλλά λειτουργούν εντελώ αποκομμένα το ένα από το άλλο. Και επομένω να μην συνεισφέρει το ένα στο έργο του άλλου. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία σφαιρική αξιολόγηση για μία Χ χώρα, για παράδειγμα, σε σχέση με το τι κάνει για την καταπολέμηση του ζητήματος αυτού και μέσω της δράσης των θεσμικών της οργάνων. Το εγχείρημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ουσιαστικά αντιστοιχεί σε ένα σύστημα αξιολόγηση ομοτήμων. Η έκθεση αυτή τελικά πηγαίνει στους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων, είναι μια έκθεση δημόσια, σε καμία περίπτωση εμπιστευτική και επομένως μπορεί οποιοδήποτε να πει «Αγια η χή χώρα τελικά δεν μας βοηθά στην καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, γιατί ενδεχομένω να εμφανίζονται στη χώρα αυτή τα φαινόμενα τα οποία έθιξε ο κύριο Στάιερ πριν από λίγο. Συνεπώς λοιπόν, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις που εμφανίζονται στη δική μας, στην αφρικανική πλευρά, να αντιμετωπίσουμε δηλαδή το ζήτημα της έλλειψης διαφάνειας και το Παράλληλα επίσης, θα πρέπει η Αφρικανική Ένωση στο σύνολό της να μπορεί να αναλάβει δράση για το ζήτημα της δημιουργίας ικανοτήτων, διοικητικών ικανοτήτων στις αφρικανικές χώρες. Μπορούμε για παράδειγμα να δούμε ότι έχουμε μία μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η οποία όμως τελικά δεν μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς. Τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή. Η ίδια η χώρα τελικά μπορεί να μην έχει τη διοικητική ικανότητα προκειμένου να βελτιωθεί ως χώρα στον τομέα της καταπολέμησης των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Και αυτό λοιπόν το ζήτημα μας απασχόλησε και το συζητήσαμε με πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς συζητώντα με εκπροσώπου τη κυβέρνηση των ΗΠΑ, μα είπαν ότι μπορούν να μα βοηθήσουν προ αυτό. Με τον ίδιο τρόπο ανταποκρίθηκε και ο ΩΣΑ. Το ίδιο πράγμα μας είπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνίων. Από πάρα πολλές πλευρές υπάρχει διάθεση υποστήριξη των Αφρικανικών κρατών ως προς τη διοικητική τους ικανότητα, η οποία όμως όπως σας εξήγησα είναι πάρα πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μέσω της έκθεσης αυτής μπορούμε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για το τι κάνουν οι αφρικανικές χώρες οι ίδιες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και όχι να κάνουν τελικά αυτό το οποίο κάναν στο παρελθόν, επαφίονται μόνο στην εξωτερική υποστήριξη, την εξωτερική βοήθεια. Βέβαια, θα πρέπει και στις άλλες υπήρους να έχουμε τα απαραίτητα παρεμφερή μέσα. Δεν ξέρουν κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Δεν ξέρω αν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπήρχε ένας αντίστοιχος μηχανισμός αποδεκτός από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής των πεσυμφωνημένων στον τομέα αυτό. Δεν ξέρω αν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Από αφρικανικής πάντως πλευράς θα προβλέπετε κάτι τέτοιο και σαφώς συμφωνώ μαζί σας ότι το ζήτημα έχει και μια έντονη πολιτική πτυχή. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα μόνο σαν τεχνικό ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με πια πολύ υψηλή ε, εμπειρογνωμοσύνη στο ζήτημα της συλλογή των φόρων, των εσόδων κτλ. Προφανώς χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά για να έχουμε αυτά αποτελέσματα χρειαζόμαστε και την κατάλληλη πολιτική ηγεσία. Κατά την άποψή μου λοιπόν, Εξίσου σημαντικό είναι να είμαστε αρκετά ανοιχτοί, διαλλακτικοί και συνεργάσιμοι στο ζήτημα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Η διαφθορά αυτή πρέπει να καταπολεμηθεί οποιαδήποτε η μορφή των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών που προκαλεί. Η διαφθορά πρέπει να καταπολεμηθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο και με οποιαδήποτε μορφή παίρνει. Αν δεν καταπολεμήσουμε διαφθορά, δεν πρόκειται να ευοδοθούν οι προσπάθειές μας. Ελπίζω ότι με την παρέμβασή μου αυτή απάντησα σε ορισμένες από τις ερωτήσεις που θέσατε. Με ρωτήσατε επίσης αν οι συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικών χωρών αν θα πρέπει να προβλέπουν συγκεκριμένε προδιαγραφές για το τι πρέπει να γίνει για την πάταξη αυτού του φαινομένου. είναι σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συγκεκριμένε ρήτρε αυτέ τι συμφωνίες. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικονομική δραστηριότητα είναι παράλληλα και κοινωνική δραστηριότητα. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την οικονομική δραστηριότητα μόνο από την οπτική γωνία του κέρδους ή της απόδοσης των επενδύσεων. Η οικονομική δραστηριότητα συνεπάγεται και κοινωνική δραστηριότητα. Επομένως, είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν αναφερόμαστε στην εξορεκτική βιομηχανία να βλέπουμε όχι μόνο τις οικονομικές αλλά και τις κοινωνικές πτυχές και επιπτώσεις των αποφάσεών μας. Θα ήταν θεμητό λοιπόν να ασχοληθούμε περισσότερο με τις διμερείς αυτές συμφωνίες και να βλέπουμε τελικά τι θα πρέπει να περιέχουν οι συμφωνίες αυτές, ποιες θα πρέπει να είναι διατάξεις τους και αν θα πρέπει να κάνουν και σαφή μνήα σε ζητήματα όπως η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Συμφωνώ και μετά όσα είπατε για τα δάση. Το συζητήσαμε και το ζήτημα αυτό. Και τα δάση, όπως και οι υπόλοιποι ε, φυσικοί πόροι, θα πρέπει να υπάρχονται σε συγκεκριμένους μηχανισμούς και συστήματα προστασίας, τα οποία θα διασφαλίζουν την χρηστή τους διαχείριση και την ορθή τους εκμετάλλευση. Επομένω, τα όσα υπόθηκαν για τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων μηχανισμών για την εξωρεκτική βιομηχανία ως προς την παρακολούθηση δηλαδή του κλάδου αυτού κτλ. Ναι, με βρίσκουν σύμφωνο και θα πρέπει να ισχύουν και για τον δασοκομικό τομέα. Ξέρετε ότι στη Λιβερία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου Ορισμένοι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή του πολέμου προέρχονταν από την παράνομη εμπορία ξυλίας. Η φυστάμενη όμως κυβέρνηση τώρα της Λιβερίας έκανε το ακόλουθο. Συνεργάζεται αυτή τη στιγμή με μία επιχείρηση η οποία είναι σε θέση να παρακολουθεί κάθε δραστηριότητα υλοτομία στη χώρα αυτή. Επομένως καταγράφουν πλέον κάθε παρτίδα ξυλίας, καταχωρούν όλα τα σχετικά στοιχεία και παρακολουθούν όλη την αλυσίδα εκμετάλλευσης από το δάσος μέχρι τον ε, τελικό αποδέκτη καταναλωτή. Κατά αυτόν τον τρόπο η Λιβερία μπορεί ακριβώς να γνωρίζει πού δραστηριοποιούνται οι υλοτόμοι, ποιο είναι το ποσοστό υλοτομίας στη χώρα και πού καταλήγει. Μέσω τέτοιων μηχανισμών μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Πολλοί αναφερθήκατε στα διαμάντια τα οποία προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις. Ανάλογα συστήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν λοιπόν και για τους πολύτιμους αυτούς λίθους και γενικότερα για τα ορυκτά, προκειμένου τα έσοδα από τις δραστηριότητες αυτές να υποφελούν τους ίδιους τους πολίτες των χωρών όπου διεξάγεται αυτή η δραστηριότητα. Η κυρία Γκόμες αναφέρθηκε σε συγκεκριμένε υποθέσεις, ότι πρέπει να ασχοληθούμε με συγκεκριμένε περιπτώσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Για παράδειγμα, στα έγγραφα του Παναμά έχουμε πλέον χειροπιαστές συγκεκριμένε υποθέσεις, υποθέσεις διαφθοράς. Βέβαια, ο Παναμάς δεν είναι ο μόνος φορολογικός παράδεισος σε αυτόν τον κόσμο, αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά. Συζητήσαμε το ζήτημα αυτό με εκπροσώπους Αμερικανικής κυβέρνησης οι οποίοι μας είπαν ότι και ορισμένε πολιτείες των ΗΠΑ μπορούν να λειτουργήσουν ή έχουν λειτουργήσει ως φορολογική παράδειση και ότι και αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Νίση Κέιμαν, οι Σεϊχέλες και πολλές άλλες περιοχές. Αυτό το οποίο όμως βλέπουμε πλέον με τα αρχεία του Παναμά είναι ότι έχουμε πλέον χειροπιαστές υποθέσεις και έχει βελτιωθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο αυτό. Μπορεί να μην γνωρίζουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή ποιοι είναι ακριβώς όλοι οι φορολογικοί παράδεισοι, παράδειση παγκοσμίω, αλλά γενικότερα οι πολίτες γνωρίζουν ότι υφίστανται η φορολογική παράδεισοι. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σα και απευθύνομαι στην κυρία Γκόμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να ασχοληθούμε με χειροπιαστέ υποθέσει. Γιατί μπορούμε να δώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένα παραδείγματα για την μορφή που παίρνει το πρόβλημα αυτό. Μα είπατε επίση ότι πρέπει να υπάρχει μεταξύ μόνο μια καλύτερη συνεργασία, μια καλύτερη διάρθρωση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική λειτουργεί ως γραμματεία μας. Αυτή, να θέλετε, το φεδικό μας, ο προϊστάμενό μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μία κάποια θεσμική διασύνδεση ανάμεσα σε εσά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη γραμματεία αυτή, έτσι ώστε να μπορούμε ακόμα και σε καθημερινή βάση να ανταλλάσσουμε πληροφορίε και να είμαστε σε επαφή. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε από κοινού να ενισχύσουμε τι προσπάθειες αυτέ που πρέπει να καταβάλουμε. Από τη δική μα την πλευρά σίγουρα θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ αν μπορούσαμε να βρούμε μια τέτοια διευθέτηση. Ενδεχομένως θα μπορούσε να ασχοληθεί συγκεκριμένα μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τη δική μα πάντω την πλευρά η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική, που έχει την έδρα της στην Αντίσα Σαμπέμπα της Αιθιοπίας, είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία και να έχουμε μια καλύτερη, πιο επικοδομητική διασύνδεση. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε λίγο και με το πρόβλημα το οποίο έθιξε η κυρία Έλλη Σλάιν, ιδίως αναφερόμενη στην υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Θεωρητικά το σύστημα φαίνεται να είναι καλό. Το αν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης αυτό πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Και θα πρέπει στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε κι εμείς να συμβάλλουμε προκειμένου ένας τέτοιος μηχανισμός να λειτουργεί τελικά αποτελεσματικά και να είναι ο κατάλληλος μηχανισμός για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Το αναφέρω αυτό γιατί έχει προκύψει το εξή ζήτημα. Βλέπουμε ότι δεν είναι πολλές οι αφρικανικές αυτές χώρες που συμμετέχουν στις διάφορες φορολογικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η φοροδιαφυγή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τις αφρικανικές χώρες να ασχοληθούν οι ίδιες με το ζήτημα της πάταξης της φοροδιαφυγής. Είπαμε λοιπόν ότι ω ομάδα υψηλού επίπεδου σχετικά με τι παράνομε χρηματοοικονομικές ροές θα ασχοληθούμε και με αυτή την πρόκληση, καλώντα όλο και περισσότερε αφρικανικέ ώρε να συνταχθούν μαζί μα. Θεωρώ ότι αυτό πραγματικά θα αποφελήσει και το δικό μα το πάνελ, αλλά και τι ίδιε τι χώρε αυτέ. Το ζήτημα λοιπόν που θίξετε και αναφέρομαι στην κυρία Σλάιν, για το τι γίνεται σε σχέση με την υποβολή εκθέσεων χώρα, και σε σχέση με τα πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούμε και τις προδιαγραφές τις οποίες χρησιμοποιούμε, αν όλα βαίνουν αισίως ή αν ένα περιθώριο βελτίωσης, νομίζω ότι με την εμπλοκή περισσότερων αφρικανικών κρατών θα είμαστε σε θέση να δούμε αν υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης και θα δούμε τι τροποποιήσεις μπορούμε να επιφέρουμε. Αναφερθήκατε επίσης και στη διάβρωση της βάσης και στη μετατόπιση των κερδών Νομίζω ότι και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη συνεργασία των απτυσσόμενων χωρών. Και βέβαια για το ζήτημα αυτό συνεργαζόμαστε πιο συγκεκριμένα με τον ΩΣΑ. Απάντησες στην ερώτησή σας. Για μετά το κοτονού. Δεν το έχουμε ακόμη συζητήσει, δεν γνωρίζω. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα αυτά τα θέματα. Ποιο είναι το όραμά μας για μετά την ε, Συμφωνία Κοτονού. Ίσως η Αφρικανική Ένωση θα ήθελε, εφόσον δεν το έχει πράξει βέβαια μέχρι τώρα, να το εξετάσει το ζήτημα. Ωστόσο, φυσικά ε, και είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολεί όλους. Αναφέρατε κάποια νούμερα τι χάνει ετησίως η Αφρική από τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Μόνο τις τελευταίες λίγες ημέρες πήραμε μία έκθεση που δείχνει ότι τα αριθμητικά αυτά στοιχεία δεν αντικατοπρίζουν καν την πραγματικότητα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν προετοιμάζαμε αυτή την έκθεση, συζητήσαμε στις αρχές ίσπραξη εσόδων τις ε, νοτιοαφρικανικές και μας ανέφεραν μια υπόθεση, την περίπτωση μιας νοτιοαφρικανικής εταιρείας που άνοιξε γραφείο στη Γενέβη. Και πήρε ε, δύο άτομα από τη Γενέβη ε, και άλλους δύο ντόπιου και τους ε, απασχολεί εκεί τέσσερα άτομα λοιπόν. Και ο ένας από αυτούς αναφέρεται ως ιδιοκτήτης της εταιρείας αυτής στην Ελβετία. Μετά το γραφείο πήγε στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Το εξέτασαν από κοντά το πιστατικό οι νοτιοαφρικανικές άρχες και είδαν ότι τελικά αυτή την ε, νοτιοαφρικανική εταιρεία δεν την είχε το ελβετικό γραφείο. Ήρθαν σε επαφή λοιπόν με τις ελβετικές αρχές. Δύο δις δολάρια έπρεπε τελικά να επιστραφούν και επιστράφησαν στην ε, Νότιο Αφρική. Από μια εταιρεία λοιπόν, βλέπετε, μέσα σε 5-6 χρόνια. Αυτό που θέλω να πω με αυτό είναι ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό για την Αφρικανική Ήπειρο, γιατί χάνουμε πάρα πολλού πόρους, πάρα πολλά χρήματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε για την εκρίζωση της ε, φτώχειας, την, ε, της Είναι πράγματι πολύ σημαντικό και συμφωνώ με το σχόλιο που έγινε και από τον κύριο Κοράου. Είπατε κύριε Κορά δεν είναι μόνο ε, αφρικανικό το πρόβλημα, σίγουρα δεν είναι. Είναι παγκόσμιο, αλλά επηρεάζει πολύ την Αφρικανική Ήπειρο και γι' αυτό θα μας ενδιέφερε ιδιαίτερως να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να έχουμε απτά αποτελέσματα. Γιατί τα αποτελέσματα αυτά σημαίνουν ότι μπορούμε να χτίσουμε ε, νοσοκομεία, σχολεία, δρόμους να ε, δημιουργήσουμε, να ε, έχουμε δηλαδή πρακτικές, θετικές πρακτικές επιπτώσεις. Δεν ξέρω, έχω απαντήσει όλες τις ερωτήσεις. Ε, ευχαριστώ. Σίγουρα έχετε απαντήσει σε ερωτήσεις, θα παρακαλέσω το προσωπικό να δώσει μια συνέχεια. Έχουμε και την ομάδα εργασίας ε, σε την Επιτροπή μας. Ε, να δώσω το λόγο στον ε, συνάδελφό μου, Λίνη Σέλση, πρόεδρο της Επιτροπής Ίσης Εκπροσώπησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΑΚΕ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Θάμπο Μπέκη για την εξαιρετική παρουσίαση και το έργο ε, της Επιτροπής που είναι ένα κομβικό έγγραφο ε, για την αντιμετώπιση ενός σοβαρότατου προβλήματος ε, το οποίο για μια ακόμη φορά βλέπει το φως της δημοσιότητας μετά τις αποκαλύψεις των εγγράφων του Παναμά. Θέλω να σας ευχαριστήσω που απαντήσατε και με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια στις ερωτήσεις ε, των συναδέλφων. Φυσικά όλοι συμφωνούμε ως προς το ότι οι παράνομες ε, χρηματοοικονομικές ροές έχουν ως άμεση επίπτωση την υπανάπτυξη. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια χώρα όταν χάνει τόσο σημαντικό όγκο ε, πόρων που θα μπορούσε, αν διατίθετο, να βοηθήσει να εφαρμοστούν οι σωστές πολιτικές. Φυσικά χρειάζονται και τα οικονομικά και τα τεχνικά μέσα για την αντιμετώπιση των παρανόμων χρηματοοικονομικών ορών. Αυτό είναι δεδομένο. Ε, επισημάναμε ένα σημείο ε, στο πλαίσιο των εγγράφων του Παναμά. Πολλοί λένε ναι πράγματι, αλλά έχουμε ε, κάποια πράγματα που είναι παράνομα και κάποια που είναι νόμιμα. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη ότι δεν θα πρέπει να μας απασχολεί μόνο τα παράνομα πράγματα. Υπάρχουν και κάποια νόμιμα πράγματα που είναι ανήθικα όμως. Και εδώ βέβαια ε, μπαίνουμε στην καρδιά του προβλήματος ε, και έχουμε και την πολιτική διάσταση. Υπάρχει η πολιτική βούληση. Αν δεν υπάρχει, και πρέπει να σας πω, και δεν ξέρω κατά πώς αυτό θα καθησυχάσει τη συνείδησή μας, ε, είχαμε πει για την Αφρικανική Διακυβέρνηση παλαιότερα και ότι δεν υπήρχε ε, παρκής αντίδραση από τις Αφρικανικές κυβερνήσεις. Δεν βλέπω αντίστοιχη βέβαια προθυμία και διάθεση ούτε από τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σήμερα. Ακούμε πολλές φορές ένα επιχείρημα ότι αφού δεν γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να το κάνουμε στη χώρα μας. Φυσικά και δεν συμφωνώ με μια τέτοια δήλωση. Η Ευρώπη είναι ένα θεσμικό δημοκρατικό κόρπους που είναι σε πολύ καλή θέση για να αποτελέσει το καλό παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο και έχει και τα μέσα η Ευρώπη να το κάνει αυτό. Μεταξύ αυτών και τα πολιτικά μέσα εφόσον εκπροσωπεί μια οικονομική ε, αγορά με πάνω από 500 εκατομμύρια φερέγγιους ε, πολίτες Άρα νομίζω ότι ε, πρέπει να δείξουμε μια πιο ενάρετη στάση, αν θέλετε. Τώρα, σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να υιοθετηθούν, όπως είπα, ενάρετες πρακτικές ε, σε πολλούς τομείς. Και αυτό που συγκρατώ ε, κατά κύριο λόγο από την δουλειά που έγινε είναι η ερώτησή σας πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν επιχειρησιακά και να λειτουργήσουν στην πράξη. Θα ήταν ενδιαφέρον, πιστεύω, να ακολουθήσουμε και τη δική σας υπόδειξη, κυρία Μακάβαν, δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε, αν θέλετε, ένα όργανο εργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της δικής σας ομάδας εργασίας και άλλων φορέων. Ένα είδος πλατφόρμας ε, που θα μπορούσε να βοηθήσει όχι μόνο τις αφρικανικές χώρες, αλλά και τις δικές μας, τις ευρωπαϊκές χώρες, ε, να έχουν την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή δυνατότητα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτές τις ροές. Αυτά ήθελα να πω. Και συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όσα υπόθηκαν, ότι σε όλο αυτό ε, το πλαίσιο θα πρέπει, φυσικά εγώ δεν λέω ότι πρέπει να αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο, γιατί είμαι υπέροχο οικονομία τη αγορά. αγοράς. Αλλά αντιλαμβάνομαι απολύτω ότι η οικονομία τη αγορά, έτσι όπως αναπτύσσεται σήμερα, δεν μπορεί ε, να επιβιώσει μακροπρόθεσμα με, αυτό το, ε, με αυτή τη μορφή. Άρα, και από πολιτική πλευρά βέβαια είναι ένα ζήτημα, το είπε και ο συνάδελφο Κοράου πάρα πολύ σωστά, ότι δηλαδή σήμερα την πολιτική εξουσία την έχουν σε μεγάλο βαθμό οικονομικέ δυνάμει, και χρηματοπιστωτικέ δυνάμει. Και πράγματι, οι χρηματοπιστωτικέ δυνάμει πολλέ φορέ χρησιμοποιούν επιχειρήματα σκανδαλώδη, όπω αυτό που έλεγα πριν, ότι αν δεν γίνεται κάτι σε παγκόσμιο δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο χώρα. Και πίσω από αυτό το επιχείρημα κρύβονται και πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτε. Πάντω, η όλη συζήτηση είναι συναρπαστική. Εδώ, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαπιστώνω ότι υπάρχει μια επιτάχυνση και θα έλεγα εκθετική και σε ό,τι αφορά την ε, συνειδητοποίηση του προβλήματος και την αναζήτηση λύσεων, αλλά είναι σημαντικό να το υπενθυμίσουμε ότι η πολιτική είναι αυτή που θα πρέπει να δώσει την όθηση. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε που είστε η πηγή που ασχολείστε συνεχώς με αυτό το ζήτημα και να μείζον κατ' ζήτημα είναι αυτοί οι μηχανισμοί που σε αιτήσια βάση αξιολογούν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους. Φυσικά πρέπει να είναι κοινή στόχη. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Μπέγκη και όλη την ομάδα του από την Αφρικανική Ένωση και θα δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Επιτροπή αυτή του κ. Μπαϊκή. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε έπειτα με το επόμενο εξίσου σημαντικό σημείο της μερίσιας διάταξης.